Αρχίζει η συνεδρίαση της Επιτροπής Προϋπολογισμών. Σύμφωνα με ε, τους κανόνες που σας ε, έδωσα την προηγούμενη εβδομάδα, θέλω να σας ενημερώσω για το τι συζήτησαν οι συντονιστές σήμερα, έτσι ώστε να το επιβεβαιώσετε κι εσείς. Πρώτα απ' όλα θα έχουμε επαφές με την Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων προκειμένου όταν φτάσει η ώρα να ετοιμάσουμε έκθεση πρωτοβουλίας για το σχέδιο επενδύσεων των 300 δισεκατομμυρίων ευρώ του Πρόεδρου Γιούγκερ. Όσον αφορά τώρα τα θέματα που έχουμε προσυζήτηση, η κυρία Ολμέγερ ορίστηκε η συγγήτρια, μάλλον συντάκτρια γνωμοδότησης για δύο εκθέσεις της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ Πρόκειται για το Smart Border Package και στη συνέχεια ζητήσαμε να εφαρμοστεί το άρθρο 55 για τις κοινέ αρμοδιότητες επιτροπών με την Υποπιτροπή Άμυνας. Προκειμένου να συντάξουμε έκθεση πρωτοβουλίας για την χρηματοδότηση αποστολών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 τις δύο τροπολογίες, διότι πιστεύω και εγώ ότι είναι πάρα πολύ καλές, τις δύο τροπολογίες της γενικής μας ε, εισηγήτριας. Μετά λοιπόν από αυτά θα ψηφίσουμε όλοι μαζί με τον ίδιο τρόπο. Ενία. Καλώς έχουμε την τροπολογία λοιπόν αριθμός 1. Υπέρ παρακαλώ. Ευχαριστώ. Κατά. Βλέπω δύο. Ευχαριστώ. Αποχές. Εγκρίθηκε. Περνάμε τώρα στο recital Δέλτα. Τη συζυγήτρια υπέρ, υπέρ, παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία αριθμός 2. Α νέο recital delta. Υπέρ εισηγήτρια, υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα το σύνολο του τροποποιημένου κειμένου με ονομαστική ψηφοφορία, ηλεκτρονική ψηφοφορία παρακαλώ. Μπορείτε να ψηφίσετε. Πέρα τη ψηφοφορίες. Δεν προλάβατε να ψηφίσετε. Ξανά λοιπόν. Ψηφίστε παρακαλώ. Δεν λειτουργεί το μηχάνημα. Λοιπόν, ξανά. Ψηφίζουμε και πάλι. Εντάξει τώρα. Μπορέσατε να ψηφίσετε όλοι. Πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 21 ψήφοι υπέρ και 3 ψήφοι κατά. Περνάμε τώρα σε διάφορες τροπολογίες για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Παράγραφος 2α, τροπολογία 2. Καλύπτεται. Παράγραφος 5, τροπολογία 3. Κατά. Ε, υπέρ παρακαλώ. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Αρχίζει η ψηφοφορία. Παράγραφος 5α, τροπολογία 3 πέρα τη φοφορίας. Εγκρίνεται. 14 ψήφοι υπέρ, 9 κατά. Τροπολογία 4 στην παράγραφο 9α νέα. Υπέρ. Συγκίτρια υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος β νέα. τροπολογία 5, υπέρ εισηγήτρια, υπέρ παρακαλώ. Κατά. Εγκρίνεται. Παράγραφος 13α, νέα, τροπολογία 6, υπέρ εισηγήτρια, υπέρ παρακαλώ. Κατά. Ούτε αποχές. Εγκρίνεται. 13β, νέα, τροπολογία 7, υπέρ, κατά εισηγήτρια, υπέρ παρακαλώ. ηλεκτρονικά, να ελέγξουμε. Μπορείτε να ψηφίσετε. Πέρα τη ψηφοφορίας. Δεν λειτουργεί. Το μηχάνημα ρωτάει ο πρόεδρος. 15 ψήφοι υπέρ, 8 κατά. Εγκρίνεται. Παράγραφος 13 γ, τροπολογία 8 καλύπτεται. 13 δέλτα νέα τροπολογία νέα καλύπτεται και εκλογική φορά ε, τροπολογία 1 υπέρ εισηγήτρια υπέρ παρακαλώ κατά αποχές εγκρίνεται. Ονομαστική ψηφοφορία τώρα στο τροποποιημένο κείμενο. Μπορείτε να ψηφίσετε. Πέρα τη ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 21 ψήφι υπέρ, κατά. Ερχόμαστε στη δεύτερη έκθεση για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, έκθεση Σαρβαμά. Ο συγγετής δεν έχει παρατηρήσεις, οπότε μπορούμε να αρχίσουμε να ψηφίζουμε τις τροπολογίες. Παράγραφος 1, τροπολογία αριθμός 2. Υπέρ ο εισηγητής. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 2α νέα, τροπολογία 3. Κατά ο εισηγητής. Υπέρ παρακαλώ. Ηλεκτρονικά θα ψηφίσουμε παρακαλώ. Ψηφίστε. πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 17 ψηφί υπέρ, 8 κατά. Παράγραφος 6α νέα, τροπολογία 4, καλύπτεται. Παράγραφος 7α νέα, τροπολογία 5, υπέρ ο συγκητής. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Μία. Παράγραφος 7β νέα. Τροπολογία 6. Υπέρ ο συγκητής υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 7 γάμα νέα. Τροπολογία 7. Υπέρ ο υπερ κατα αποχες εγκρινεται παραγραφος 7 γαμα νεα τροπολογια 7 υπερ ο υπέρ. υπερ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 8, τροπολογία 8, υπέρ ο εισηγητής. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δέλτα Α νέα αιτιολογική αναφορά. Τροπολογία 1 του εισηγητή υπέρ. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές δεν υπάρχουν. Και έτσι θα ψηφίσουμε τώρα το σύνολο του τροποποιημένου κειμένου με ονομαστική ψηφοφορία, ηλεκτρονική δηλαδή. Μπορείτε να ψηφίσετε. Πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. 21 ψήφοι υπέρ, 4 κατά. Περνάμε στο τμήμα 3. Βάσει της ψηφοφορίας που κάναμε, τώρα θα περάσουμε στη μεταφορά της τόσεων που είναι αναγκαίες μετά τα όσα ψηφίσαμε. Για πείτε μας λοιπόν, για τρία θέματα έχετε να μας μιλήσετε. Ίσως μπορείτε να μας μιλήσετε και για τα τρία μαζί και να ψηφίσουμε μαζί. Πρόεδρε, για τα δύο πρώτα μπορούμε μαζί, για το 26 δηλαδή και το 28. Μπορούμε να τα ψηφίσουμε μαζί. Διότι είναι αναγκαίο να ψηφίσουμε τις δύο αυτές προτάσεις εφόσον επιτρέπουν να είναι η πράξη αυτά που μόλις ψηφίσαμε, γιατί έτσι θα μεταφερθούν οι πιστώσεις που βρίσκονται στο αποθεματικό του Ευρωπαϊκού Ταμείου για την Παγκοσμιοποίηση στο ίδιο το Ταμείο. Και έτσι τα χρήματα αυτά θα μπορέσουν να εκταμιευθούν. Ζητάω λοιπόν να υπερψηφίσουμε τα δύο αυτά αιτήματα. Ωραία, λέει ο Πρόεδρος. Ποιοι είναι υπέρ, παρακαλώ. Κατά. Κατά. Αποχές. Οι τροπολογίες 26 28 εγκρίνονται. Τροπολογία 31 τώρα. Για την τροπολογία αυτή, λέει ο κύριο Ντεπρέ, τα πράγματα είναι κάπω διαφορετικά. Κάθε χρόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοιμάζει μία πρόταση που είναι, ονομάζεται ε, συνολική μεταφορά που επιτρέπει να υπάρξει νέα ισορροπία στις πληρωμές για το τρέχον έτος. Κατά τη διάρκεια λοιπόν του έτους, οι χρηματοδοτήσεις από διάφορες γραμμές ικανοποιούνται όσο γίνεται περισσότερο με εσωτερικές μεταφορές στα πλαίσια του ίδιου του κεφαλαίου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να το κάνει αυτό, προβλέπεται εξάλλου από τον δημοσιονομικό κανονισμό. Όμως, όταν είμαστε εκτός των ε, κεφαλαίων αυτών, χρειάζεται η ειδική άδεια. Και αυτό ακριβώς τώρα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δηλαδή, η πρόταση μεταφοράς έχει να κάνει με ανάγκες πιστώσεων που δεν μπορούν να καλυφθούν από εσωτερικές μεταφορές από το ίδιο το κεφάλαιο. Πρόκειται για το 2014 για πληρωμές 475,1 εκατομμυρίων. 25% περίπου των πληρωμών που επιτρέπονται από τον προπολογισμό του 2014. Αν θέλετε μπορώ να σας δώσω περισσότερες λεπτομέρειες αν κάποιος ενδιαφέρεται. Πρόκειται, αν θέλετε να σας εξηγήσω, θα μας πάρει βέβαια 20 λεπτά περίπου, αλλά νομίζω ότι το ίδιο το κείμενο της Επιτροπής και τόσα σας είπα. Ελπίζω να σας πείθουν για την συνολική αυτή πληρωμή. Δεν βλέπω να έχει κανείς αντιρρήσεις, λέει ο Πρόεδρος. Πρόκειται για ένα μέτρο το οποίο διασφαλίζει τις πληρωμές, έτσι δεν είναι, σύμφωνα με τους κανόνες. Και να μην υπάρχουν έτσι χρέη, γιατί καμιά φορά σε κάποιες γραμμές δεν χρησιμοποιούνται οι πιστώσεις, ενώ χρειάζονται κάπου αλλού και εκεί δεν υπάρχουν επιστώσει. Να λοιπόν ένα μέτρο μεταφορά που επιτρέπει να επιταχύνονται οι πληρωμέ. Ψηφίζουμε λοιπόν την τροπολογία αριθμό 31. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Ένας αποχές. Η τροπολογία 31 εγκρίνεται συνεπώς. Κυρία Χολμέγερ. Α, έχετε κι άλλα. Κύριε Ντεπρέ. Πρόκειται για το άρθρο 50 για αλλαγή θέσης. Έχετε το λόγο. Πρόεδρε, είναι πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εδώ ακούστε με παρακαλώ. Και αν καταλάβετε τίποτα, μου λέτε, λέει ο κύριος Ντεπρέ. Στόχο έχει η πρόταση αυτή 45 θέσεις AST3 μονίμου προσωπικού, μια θέση AST4 και 26 θέσεις προσωρινών υπαλλήλων να γίνουν ASTS, 10 θέσεις προσωρινών να γίνουν AST4 και νέα θέσεις προσωρινών προσωρινών 3. Αυτές να γίνουν AST ES 4, όλες μαζί και 45. Όσον αφορά την Όλαφ, για να τα πω όλα, υπάρχει το αίτημα επίσης αλλαγής από από 2 θέσεων να γίνουν AST 1 Όποιος μετά από μένα μπορεί να τα επαναλάβει όλα αυτά, σίγουρα διανοητικά θα είναι πολύ δυνατός, λέει ο κύριος Ντεπρέ. Βάσει του άρθρου 50 λοιπόν του Δημοσιονομικού Κανονισμού, η Επιτροπή Προπολογισμών έχει τρει εβδομάδε στη διάθεσή τη για να προφέρει ένσταση. Έχουμε δηλαδή στη διάθεσή μα μέχρι τι 27 Οκτωβρίου. Αν δεν υπάρξει ένσταση μέχρι τότε, τότε η μεταφορά αυτή αρχίζει να ισχύει χωρί να χρειάζεται να γίνει ψηφοφορία επίσημα. Εδώ πέρα υπάρχουν όμως δύο ερωτήσεις. Πρώτον, γιατί γίνονται όλα αυτά. Εγώ είδα ένα εγγραφό στο οποίο εξηγεί ότι είναι για να δημιουργηθεί καλύτερα το γραφείο της Νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής η συνεργασία των ε, επιτρόπων δηλαδή. Απ' την άλλη μεριά δημοσιονομικά πρέπει να είναι ουδέτερη η πρόταση. Και εδώ βλέπω ότι οι δαπάνες θα είναι λιγότερες, αν τουλάχιστον καταλαβαίνω καλά τον πίνακα που έχω μπροστά μου. Πράγμα που σημαίνει ότι κατά, πο... κατά πάσα πιθανότητα οι θέσεις αυτές υποβιβάζονται. Εγώ δεν τα καταλαβαίνω λοιπόν όλα αυτά. Ας μου τα εξηγήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλιώς εγώ προτείνω ένσταση από την πλευρά μας γιατί δεν καταλαβαίνω ούτε γιατί χρειάζεται αυτό, ούτε γιατί γίνεται ο υποβιβασμός αυτός. Θα ήθελε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Και άρα... Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν μπορεί να μας εξηγήσει, βεβαίως. Πολύ θα ήθελα. Γιατί τα έγγραφα που έχουμε στη διάθεσή μας δεν μας εξηγούν καλά. Η επιχειρηματολογία μου φαίνεται πολύ αδύναμη και δεν βλέπω καν την ουδετερότητα αυτή στον προπολογισμό. Η Επιτροπή λοιπόν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου να προσπαθήσω να εξηγήσω. Από 1η Ιανουαρίου φέτος υπάρχει μια νέα θέση στους βοηθούς βάσει των γραμματιών που έχουν δημιουργηθεί και που δεν υπήρχαν πριν. Προβλέπονται λοιπόν προσλήψεις για την γραμματιακή αυτή στήριξη σε χαμηλότερο επίπεδο, άρα και το κόστος θα είναι χαμηλότερο. Για να υλοποιηθεί αυτό η πρόταση της Επιτροπής για να μπορέσει να προσλάβει άτομα, ε, πρέπει στον κατάλογο των θέσεων να αναφέρονται οι λεπτομέρειες της κάθε θέσης ανακατηγορία και να υπάρξει εκεί μια τροποποίηση. Όταν ε, λοιπόν υπέβαλε την πρόταση προπολογισμού 2014 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν υπήρχαν αυτές οι θέσεις, δεν προβλέπονταν αυτή η γραμματεία. Τώρα στα πλαίσια του προπολογισμού 2015 ξαναβλέπουμε λοιπόν τον πίνακα και προσπαθούμε να τον προσαρμόσουμε στις νέες κατηγορίες καθηκόντων, λαμβάνοντας υπόψη τη δημιουργία αυτής της γραμματείας δηλαδή. Τώρα είμαστε στα τέλη μιας χρονιάς εκεί που υπάρχουν κενές θέσεις μπορούμε να προσλάβουμε σε χαμηλότερο επίπεδο υπαλλήλους για να καλύψουμε τις ανάγκες της γραμματείας, για ορισμένους επιτρόπους, για παράδειγμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι διατεθειμένη λοιπόν να προσλάβει νέο προσωπικό, αλλά η περιγραφή που έχουμε για τις συγκεκριμένες θέσεις μέχρι τώρα δεν ανταποκρίνεται. Γι' αυτό και πρέπει να βασιστούμε στο άρθρο 50 που προβλέπει ευελιξία των κριτηρίων ώστε να μπορέσουμε ήδη να προσλάβουμε προσωπικό για τις γραμματιακές ανάγκες για τους δύο τελευταίους αυτούς μήνες της χρονιάς. Πρέπει να δοθεί η άδεια. Και κάνουμε και κάποιες οικονομίες, για δύο μήνες βέβαια. Στη συνέχεια με τον προπολογισμό 2015 ήδη προβλέπεται η νέα δομή και ο αριθμός θέσεων που χρειάζεται και τα νούμερα τα αποκρίνονται όπως πρέπει. Ωραία. Σε ένα βαθμό καταλάβαμε. Κύριε Ντεπρέ, άκουσα πολύ ενδιαφέρον τα όσα είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά ειλικρινά αναρωτιέμαι γιατί δεν μπορούν όλα αυτά να μας τα εξηγήσουν ε, ξεκάθαρα. Να μας πούνε για ποια θέση, για τι καθήκοντα, για ποιον επίτροπο, γιατί λειτουργούν οι υπηρεσίες των επιτρόπων, έτσι δεν είναι. Οπότε γιατί πρέπει να περάσουμε από όλα αυτά. Δεν ξέρω, ο καθένας σας κρίνει όπως νομίζει εδώ. Εγώ προσωπικά δεν είμαι διατεθειμένος να δεχτώ την πρόταση αυτή και προτείνω να αναβληθεί η απόφαση. Ο κύριος ε, Ναλή. Πρόεδρε, νομίζω ότι προφανώς δεν είναι ξεκάθαρο. Γιατί τι γίνεται με το ήδη υπάρχον προσωπικό. Εγώ νομίζω ότι χρειαζόμαστε περισσότερες πληροφορίες πριν να αποφασίσουμε. Στηρίζω λοιπόν αυτό που προτείνει ο κύριος Δεπρέ. Δεν με ικανοποίησαν ούτε οι εξηγήσει που μας έδωσε πριν από λίγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρόεδρος, προτείνω να ψηφίσουμε αυτό που ζήτησε ο εισηγητής, την αναβολή δηλαδή της απόφασης, ώστε να μπορέσουμε έτσι να ζητήσουμε περισσότερες πληροφορίες. Ποιοι συμφωνούν με τον εισηγητή για την αναβολή αυτή λοιπόν. Κατά. Αποχές. Έχουμε κάποιες αποχές. Κανείς κατά όμως. Ωραία, η πλειοψηφία ζητάει περισσότερες πληροφορίες. Κύριε Πρεζά, κάνατε ό,τι μπορούσατε, αλλά θα επανέλθετε στην επόμενη συνεδρίασή μας να μας τα εξηγήσετε καλύτερα. Η κυρία Ολμέγερ δεν έχει έρθει, έχει ανελημμένες υποχρεώσεις αλλού. Ο κύριος Φερνάντες όμως ίσως θα μπορούσε να αντικαταστήσει την εισηγήτρια. Κύριε Φερνάντες. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω πορτογαλικά. Έχουμε δύο προτάσεις που αφορούν το δικαστήριο. Η μία μεταφορά αφορά 897.000 ευρώ και πρόκειται για μισθολογική προσαρμογή, είναι υποχρέωση, νομική υποχρέωση και η δεύτερη μεταφορά αφορά 413.000 ευρώ και έχει να κάνει με τη χρηματοδότηση ηλεκτρονικών δημοσιεύσεων. Δεν υπάρχει πρόβλημα για την έγκριση αυτών των δύο μεταφορών να σας παρουσιάσω ήδη μια αλλαγή που αφορά την Επιτροπή των Περιφερειών και την μετατροπή θέσεων που έχει επίσης μια ουδέτερη ε, δημοσιονομική επίπτωση. Είμαι υπέρ λοιπόν των τριών αυτών περιπτώσεων μεταφορών. Ευχαριστώ. Ίσως μπορούμε να ψηφίσουμε unblock για τις τρεις αυτές μεταφορές. Ψηφίζουμε λοιπόν ποιοι είναι υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. Τελειώσαμε λοιπόν με τις ψηφοφορίες. Και τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Φερνάντες για να μας παρουσιάσει την έκθεσή του για την ε, αλληλευτική συμφωνία με την ε, δημοκρατία του Σαοτομέ και Πρίνσιπε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρόκειται για ένα αλληλευτικό πρωτόκολλο συμφωνία που αφορά ε, τα αλληλευτικά δικαιώματα με μία ε, οικονομική ε, αντιστάθμιση. Πρόκειται για μια συμφωνία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Δημοκρατία του Σαοτομέ και Πρίνσιπε ε, και για μια διάρκεια τεσσάρων ετών και για ένα ποσό 2.805.000 ευρώ. Μισά-μισά περίπου για το πρώτο έτος και πρόκειται για 7.000 τόνους ετησίως. στηρίζεται η τομεακή ε, αλληλεία στο Σάοτομε και Πρίνσιπε, δηλαδή η ρεστεχνική και μικρής κλίμακας ε, αλληλεία ο έλεγχος και η καταπολέμηση της παράνομης αλληλείας, τα ευρωπαϊκά ε, σκάφη μπορούν να αλλιεύουν εκεί. Πρόκειται για 55 ε, ευρώ ε, τον τόνο που αυξάνεται η ευρωπαϊκή ενίσχυση και 50 ευρώ το χρόνο από το, για τον τέταρτο χρόνο. Καλύπτονται επίσης ε, όλα τα θέματα τα περιβαλλοντικά και προστασίας ε, των βυθών. Γι' αυτό και δεν βλέπω να υπάρχει καμία αντίρρηση για την έγκριση αυτού του αλευτικού πρωτοκόλου. Σας ευχαριστώ κύριε Φερνάντες. Θα ήθελε κάποιος να πάρει το λόγο για αυτή την έκθεση. Όχι. Να θυμίσω ότι οι σχετικές τροπολογίες θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι στις 23 Οκτωβρίου, ότι η ψηφοφορία στην Επιτροπή Προϋπολογισμού θα γίνει στις 20 Νοεμβρίου, στην Επιτροπή Αλληλείας 3 Δεκεμβρίου και οι διατάξεις αυτές θα υποβληθούν στην Ολομέλεια τον Ιανουάριο. Τώρα θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Στεφανέκ, για την έκθεση περί κινητοποίησης του Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση έκθεση σχετικά με την Άντερσεν της Ιρλανδίας. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε η Ιρλανδία υπέβαλε μια αίτηση για χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση μετά από 171 απολύσεις στην εταιρεία από την εταιρεία Andersen, η οποία κατασκεύαζε ε, κοσμήματα. Αυτή η υπόθεση ε, αφορά μια, την περίοδο από τον Οκτώβριο του 2013 μέχρι το Φεβρουάριο του 2014. Πρόκειται για 171 ανθρώπους, σχεδόν το 70% αυτών είναι ε, γυναίκες οι οποίες έμειναν άνεργες. Συνολική συμβολή, συνεισφορά που προτείνεται είναι 1,5 εκατομμύριο ευρώ το οποίο συνδέεται με βασικές ε, μεταρρυθμίσεις ε, στο χώρο εργασίας λόγω της παγκοσμιοποίησης. Εγώ προτείνω ε, ότι αυτή η πρόταση δεν καλύπτει το κατόφλι των 300 εργαζομένων, όμως λόγω εξαιρετικών περιστάσεων και η Κομισιόν υποστηρίζει την υπόθεση αυτή και γι' αυτό και εγώ με τη σειρά μου υποστηρίζω την έγκριση αυτής της πρότασης. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Υπάρχουν εδώ ε, παρεμβάσεις. Θέλει κανείς να πάρει το λόγο για την έκθεση του κυρίου Στεφανέκ. Να πω ότι οι τροπολογίες μπορούν να κατατεθούν μέχρι τις 16 Οκτωβρίου. Όχι, στις 16 Οκτωβρίου θα εξεταστεί ε, το θέμα από την Επιτροπή Απασχόλησης. 23 Δεκεμβρίου Οκτωβρίου μάλλον, ε, στις 12 το μεσημέρι είναι η προθεσμία για υποβολή τροπολογιών. 3 και 4 Νοεμβρίου θα ψηφιστεί στην Επιτροπή Προπολογισμού και επίσης τον Νοέμβριο θα υιοθετηθεί το κείμενο από την Ολομέλεια. Τώρα το λόγο έχει ο κύριος Νεγκρέσκου για την έκθεση που αφορά το Sprinter Stores. Πρόκειται για ένα αίτημα από πλευράς των ελληνικών αρχών για την κινητοποίηση του Ταμείου ε, για την Παγκοσμιοποίηση μετά από την απόλυση ε, πολλών εργαζομένων σε αυτή την εταιρεία Spinder Stores η οποία κήρυξε πτώχευση. Πρόκειται για... ...761 ανθρώπους που απολύθηκαν. Ήταν μια πολύ δραστήρια εταιρεία και η οποία επλήγει πολύ σοβαρά στη διάρκεια της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα. Με βάση τα στοιχεία που έχουμε στη διαθεσή μας, η Ελλάδα εδώ και έξι χρόνια διανύει μια πολύ σοβαρή ύφεση, ύφεση η οποία έχει οδηγήσει σε πολλές απολύσεις και σε πολύ μεγάλη μείωση της ε, κατανάλωσης. Αυτή η εταιρεία ήταν μια από τις πιο σημαντικές στον τομέα της ένδυσης στην Ελλάδα, με πάνω από 1.500 εργαζόμενους και πτώχευσε λόγω της οικονομικής κρίσης. Όσον αφορά λοιπόν αυτό το αίτημα κινητοποίηση του Ταμείου ε, Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση, τα κριτήρια πληρούνται. Πρόκειται για ένα ε, σχέδιο που αφορά 12 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 11.900 ε, στοχεύουν σε συγκεκριμένες δράσεις, ενώ το Ταμείο Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση θα πρέπει να αποταμιεύσει 7.290.000 ευρώ. Πρόκειται δηλαδή για συμμετοχή 60%. Έχουν τηρηθεί οι προθεσμίες ε, όσον αφορά την ισότητα ευκαιριών, την ε, έλευση διακρίσεων. Υποστηρίζω λοιπόν αυτό το αίτημα και οι συνάδελφοι που θέλουν να καταθέσουν ε, τροπολογίες φυσικά ε, είναι ευπρόσδεκτοι. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Σιγητά. Υπάρχουν ερωτήσεις, παρατηρήσεις, όχι. Λοιπόν, να σας πω τότε ότι η Επιτροπή Απασχόλησης θα εξετάσει το θέμα στις 16 του μηνός. Στις 23 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι είναι η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών για την έκθεση που μόλις μας ε, παρουσιάσατε. 3 και 4 Νοεμβρίου θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή Προϋπολογισμού και η Ολομέλεια θα ε, ε, ψηφίσει για το κείμενο στην Σύνοδο του Νοεμβρίου. Πριν να περάσουμε στις συνεδρίαση και κλεισμένο των θυρών, θα ήθελα τώρα να εξετάσουμε την έκθεση που αφορά την κτηριακή πολιτική. Η κυρία Χολμάιερ δεν είναι σήμερα διαθέσιμη για να μας παρουσιάσει την έκθεση αυτή. Ίσως ο κύριος Φερνάντες να μπορούσε να μας ε, ενημερώσει για την κτηριακή πολιτική. Την έκθεση της κυρίας Χολμάγερ που απουσιάζει. Μάλιστα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για το θέμα Τη Κένιας και την πρεσβεία στο Ναϊρόμπι. Θα τα πω στα πορτοκαλικά καλύτερα. η εισηγήτριά μας ζητά πιο λεπτομερείς ε, πληροφορίες για το θέμα και επί τη βάση του άρθρου 203 του Δημοσιονομικού Κανονισμού προτείνει ε, για να έχουμε καλύτερη ανάλυση και να σχηματίσουμε σωστότερη γνώμη να δοθεί μία παράταση της προθεσμίας κατά δύο εβδομάδες ώστε να μπορέσουμε να εκφραστούμε για αυτό το θέμα. Ακριβώς αυτό προτείνει η εισηγήτριά μας. Και εγώ συμφωνώ και ζητά μάλλον τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής μας. Παράταση για δύο εβδομάδες για την εξέταση αυτού του θέματος. Μάλιστα, δεν υπάρχει αντίρρηση. Θα αναβάλουμε κατά δύο εβδομάδες ε, την εξέταση αυτού του θέματος. κυρία Χολμάγερ θα έρθει για να μας ενημερώσει για τη γνώμη της. Άρα λοιπόν θα έχουμε και πάλι το θέμα αυτό στην ημερησία διάταξη. Αυτά λοιπόν ολοκληρώθηκε τώρα η δημόσια συνεδρίαση και θα περάσουμε στην συνεδρίαση και κλεισμένων των θυρών. Διακόπτουμε για τρία λεπτά έτσι ώστε οι μη έχοντες εργασία να εξέλθουν τις αιθούσεις. Ne reste ici que les représentants du Parlement.